δεύτερη ανακοίνωση είναι ότι ενημέρωσε ο πρόεδρος χθες ε, ε, σε σχέση με κάποιες αποφάσεις Επιτροπής Θερματικών Υποθέσεων και θεωρούνται και οι συστάσεις αυτές ότι εγκρίνονται. με το άρθρο